έχω πάρει όρκο ε, στο Πολωνικό Σύνταγμα όταν ξεκίνησα τη δουλειά μου και προσπαθώ να παραμείνω έντιμος σε ό,τι αφορά τον όρκο αυτό και να προσπίσω τα συμφέροντα των Πολωνών πολιτών. Για μένα αυτό πραγματικά εμπεριέχει τους ανθρώπους τους οποίους καλούμαστε να υπερασπιστούμε σε τέτοιες καταστάσεις. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που προασπίζονται το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία μας και πραγματικά αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της δημοκρατίας μας, των συστημάτων από τα οποία όλοι μας ωφελούμαστε. Οι εισαγγελείς λοιπόν αυτοί, αυτοί οι δικηγόροι είναι και οι δικαστές είναι μέλη αυτού του τριμερού συστήματος, το οποίο έχει τεθεί σε εφαρμογή για να προστατεύσει τη δημοκρατία μας και όντως, όπως είπαν οι συνάδελφοι, αυτά που βλέπουμε στην Πολωνία τα τελευταία χρόνια είναι μια εναρχιστρωμένη εκστρατεία κατά αυτής της πολύ σημαντικής ραχοκοκαλιάς και το είπε, ανέφερε τις σχετικές εξελίξεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο Κοινοβούλιο έχουμε λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να προσπίσουμε το κράτος δικαίου και τους Ευρωπαίους πολίτες και τους Πολωνούς πολίτες. Αλλά πιστεύω ότι η διαδικασία από το άρθρο 7 έχει συχνά αποδειχθεί ότι δεν είναι αρκετά γρήγορη και δεν είναι αρκετά ευέλικτη για να αντιμετωπίσει τα θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσει. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν μια συνολική λύση. Και ο μηχανισμός κράτους δικαίου είναι ένα από τα εργαλεία που χρειαζόμαστε μαζί με τα θέματα και τις κυρώσεις στο, τα μέτρα προπολογισμού και χρηματοδότηση. Και θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι ελπίζω πραγματικά η κρατική Προεδρία να αποτελέσει υπόδειγμα για να προσπιστεί το κράτος δικαίου. Αλλά ό,τι και να συμβεί, να έχετε υπόψη σας ότι το κοινοβούλιο αυτό θα συνεχίσει να υπερασπίζεται το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μάντισον. Σας ευχαριστώ. Αυτή τη, στιγμή θα Αυτή τη φορά θα μιλήσω εστονικά. Καταρχήν θα ήθελα να ευχηθώ καλή δύναμη και καλό κουράγιο στους Πολωνούς συναδέλφους. Ελπίζω να επιβιώσετε. Και θα ήθελα να μάθω, οι Πολωνοί δικαστές με τους οποίους μιλήσατε και αυτός που είπε ότι ορκίστηκε στο Σύνταγμα να προστατεύσει τη δικαστική τάξη στην Πολωνία, πότε έδωσε τον όρκο, μήπως επί Σοβιετικού καθεστώτος, μήπως όταν η Πολωνία ήταν υπό την κατοχή ε, της Σοβιετικής Ένωσης. Γιατί αν τότε έδωσε τον όρκο δεν χρειάζεται να τον τηρήσει, γιατί τότε δεν εργαζόταν για την Πολωνία ο άνθρωπος αυτό, αλλά για το κομμουνιστικό καθεστώς θα μπορούσατε να πείτε ότι είναι έσχος, αλλά θα πρέπει να διδαχτούμε από την ιστορία. Πριν από 30 μήνε είχαμε εκλογέ στην Πολωνία και 43% του πολωνικού εκλογικού σώματο ψήφισε το συντηρητικό πολωνικό κόμμα. 43% αυτό είναι γεγονό. Είναι πολύ ισχυρή η δημοκρατική εντολή τη πολωνική κυβέρνηση για τη διεξαγωγή μεταρρυθμίσεων. Επίση, μιλήσατε για αρχέ και αξίε και το κράτο δικαίου. Μην με διακόπτετε. Τώρα σιωπή. Θα μιλήσετε αργότερα. Πριν από λίγο μιλήσαμε για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και πολλοί ομιλητές, πολλοί συνάδελφοι είχαν μιλήσει υπέρ του κόκκινου στρατού που, που έσωσε τάχα τον κόσμο αυτό συνάδει με τις ευρωπαϊκές αξίες, δηλαδή επενείται το καθεστώς που δολοφόνησε στο Κατίν 20.000 Πολωνούς αξιωματικούς. Αυτό συνάδει με τις ευρωπαϊκές αξίες. Για σκεφτείτε το παρακαλώ. Έχω μία μπλε κάρτα. Την δέχεστε, κύριε Μάντισον, φυσικά. Έχετε μπλε κάρτα, παρακαλώ, συνάδελφε. σας παρακαλέσω το εξής και όλοι όσοι το άκουσαν δεν μπορούν να περιμένουν ε, την επόμενο θέμα που θα συζητήσουμε με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος ε, μετά από την ε, απόφαση του δικαστηρίου ήταν, αποκαλύφθηκε ότι ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος και συμβάλλει στη μη επίλυση των προβλημάτων με την Πολωνία. Μπορείτε λοιπόν να περιμένετε και μπορείτε φυσικά να πάρετε το λόγο από αυτού. αν δεν ήσταν ε, από την αρχή στη συζήτηση, μην προσπαθείτε με, το, με την μπλε κάρτα να αυξήσετε το χρόνο αγόρευσή σας, αλλά καλή ιδέα, θα το έχω υπόψη στο μέλλον. Επόμενη ομιλητρία. Η κυρία Μπέατα Σίντουο, ε, Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Οι δικαστές στην Πολωνία είναι ελεύθεροι και ανεξάρτητοι. Η Πολωνία είναι μια χώρα με κράτος δικαίου, με ευνομία. Ε, κάθε, κάθε συνάδελφος που ισχυρίζεται το αντίθετο λέει ψέματα. Αυτό το γνωρίζουν όλοι οι Πολωνοί που βρίσκονται στην αίθουσα, ακόμη και οι δικαστές που έχετε προσκαλέσει. Για τέσσερις, τέσσερα χρόνια, τότε που είχαμε την άδοξη αυτή επέτειο της, των συναδέλφων, τον, είχα την τιμή ως Πολωνή να εκπροσωπήσω την πατρίδα μου εδώ στην συζήτηση που είχαμε ε, για την Ευρώπη στο Στρασβούργο. Τότε Είχαμε μιλήσει για την κατάσταση στην Πολωνία, για τις μεταρρυθμίσεις, για το τι χρειάζεται να γίνει στην Πολωνία. Και μάλιστα οι πολίτες μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους, έδωσαν την ψήφο τους στο κόμμα νόμος και δικαιοσύνη και για τα τέσσερα τελευταία χρόνια εφαρμόσαμε πολλές μεταρρυθμίσεις, κοινωνικές, οικονομικές, διοικητικές. Αυτό το εκτίμησαν οι Πολωνοί πολίτες και μας έδωσαν εκ νέου την εμπιστοσύνη τους και πάλι μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη και την ψήφο τους για να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις που είχαμε ξεκινήσει και μέσα σε αυτά τα τέσσερα χρόνια κάναμε πολλά καλά. Αλλά οι Πολωνοί εξακολουθούν να περιμένουν από εμά να ολοκληρώσουμε τις μεταρρυθμίσεις, να ολοκληρώσουμε και τη μεταρρύθμιση στη δικαστική εξουσία. Γιατί η δικαιοσύνη, η δικαστική εξουσία θα πρέπει να υπηρετεί τους πολίτες και να μην προστατεύει συγκεκριμένα προνόμια που θέλουν να διαφυλάξουν οι ομάδες, οι συγκεκριμένες ομάδες. Επανειλημμένος η πολωνική κυβέρνηση και μάλιστα και εγώ εδώ μπροστά σας πριν από τέσσερα χρόνια, όταν ήμουν πρωθυπουργό, σας εξήγησα πόσο απαραίτητε είναι στην Πολωνία οι μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό σύστημα. Γιατί η δικαιοσύνη ήταν ε, η ο μόνος θεσμός που δεν έχει μεταρρυθμιστεί μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος και είναι το μόνο απομεινάρι ε, του κομμουνισμού σε μερικές χώρες. Και το γνωρίζει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το γνωρίζουν και πολλοί ευρωβουλευτέ, γιατί το έχουμε συζητήσει επανειλημμένω. Και γι' αυτό ξεκινήσαμε τι σχετικέ μεταρρυθμίσει στη δικαιοσύνη. Και μάλιστα οι μεταρρυθμίσει αυτέ είναι συνταγματικέ, συνάδουν με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο, αλλά περισσότερο από όλα συνάδουν με την βούληση του πολωνικού λαού, γιατί αυτήν υπηρετούμε. Ήμασταν ανέκαθεν ανοιχτοί στο διάλογο και ήμασταν ανέκαθεν πρόθυμοι να δώσουμε διευκρινίσεις και εξηγήσεις. Για να γίνει όμως διάλογος χρειάζονται δύο συνομιλητές και θα πρέπει να είναι ανοιχτή στο διάλογο και δεν φαίνεται να υπάρχει αυτό. Δυστυχώς ο πρόεδρος διακόπτει το μικρόφωνο της ομιλήτριας. Θα ήθελα να επενθυμίσω τους κανόνες και να τηρήσω τους κανόνες που έθεσε ο προηγούμενος πρόεδρος. Αναομιλητή μόνο μία μπλε κάρτα και καμία μπλε κάρτα από άτομα τα οποία είναι ήδη στον κατάλογο των ομιλητών. Γι' αυτό λοιπόν να παρακαλέσω τον κ. Τσικόρσκι να κάνει την ερώτησή του. Ευχαριστώ. Η πρώην Πρωθυπουργό Σίντουο ε, μα διαβεβαίωσε ότι όλα όσα γίνονται στην Πολωνία είναι συμβατά με το Σύνταγμα. Δεν το γνωρίζουμε όμω αυτό, γιατί η Πρωθυπουργό Σίντουο έδωσε σύσταση να μην δημοσιεύονται οι αποφάσει του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Και τότε ξεκίνησε η παραβίαση του Πολωνικού Συντάγματο και η παραβίαση τη ε, ε, ένομη τάξη τη Πολωνία. Δηλαδή, είναι μεροληπτική η πρώην Πρωθυπουργός Σίντουο στις δηλώσεις της. Είχαμε 26 ακροάσεις ε, του Σεμπάστιαν Κά, οπότε θα πρότεινα ε, τους ε, εκπροσώπους της κυβέρνησης να προσέχουν όταν μιλούν για μη παραβίαση του συντάγματος, γιατί δεν ισχύει αυτό. Η μπλε κάρτα έχει νόημα να κάνετε μια ερώτηση όχι για να συμμετέχετε στη συζήτηση. Λυπάμαι. Επόμενο ομιλητή, ο κύριο Αρβανιτή. Ναι, γιατί τι απάντησε, αυτό δεν κάνετε ερώτηση. Δεν ήταν ερώτηση, αλλά ο κύριο Σικόρσκι ε, είπε κάποια ψέματα και θα μπορούσα να τον πάω στο δικαστήριο. Γιατί δεν έχω καμία εκρεμή δίκης βάρος μου κύριε Σικώσκη. Εσείς είστε ψεύτης και ανάξιος της ε, βουλευτικής εντολής σας. Συνάδελφοι, σας παρακαλώ να προσέχετε παρακαλώ με τέτοιου είδους δηλώσεις και αιτιάσεις. Γι' αυτό γίνεται λοιπόν η συζήτηση εδώ σήμερα για το κρατός δικαίου στην Πολωνία. Αυτό είναι το θέμα και την εισαγωγή την ε, έκανε ήδη η κυρία Επίτροπος. Επόμενος ο μιλητής, ο κύριος Χαλίτσκι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από την ε, Ελλάδα είμαι και εκπροσωπώ την Γκουεντζιαρ την ε, γκουεντζιέλ την αριστερά. αν και είμαστε επιφυλακτικοί με τι παρεμβάσει της Ευρωπαϊκή ένωσης σε κράτη μέλη καθώ έχουμε πικρή εμπειρία εμεί στην ελλάδα με τα μνημόνια και με την τρόικα στη συγκεκριμένη περίπτωση της Πολωνία, συμφωνώ και συμφωνούμε σαν ομάδα με τη σύνταξη προσωρινή έκθεση που θα αφορά όχι μόνο το δικαστικό σύστημα αλλά και, και όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα που βρίσκονται σε κρίση τη στιγμή αυτή που μιλάμε. αυτή ήταν εξ αρχής η θέση της ομάδας μας αλλά και ολόκληρου του προοδευτικού τόξου όπως ακούσατε εδώ. στην πολωνία αυτή τη στιγμή υποβιβάζεται το σύνολό της, η δικαστική εξουσία προς όφελος της εκτελεστικής. βρίσκεται υποκίνδυνο η ανεξαρτησία των δικαστών τους ακούσαμε σήμερα. σκοπεύουν να καταργήσουν παράνομη ακόμα και την προσφυγή στο ευρωπαϊκό δικαστήριο στεκόμαστε δίπλα στους δικαστές στη συγκεκριμένη τους μάχη όπως και αυτοί πρέπει να είναι αλληλέγγυοι στο δίκαιο των ευάλωτων ομάδων για την ελευθερία του τύπου για το δικαίωμα του συνέρχεστε του συνεταιρίζεστε των εργαζομένων των δικαιωμάτων των γυναικών των ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο. αυτή την ευρώπη θέλουμε. αυτή την ευρώπη θέλουμε και όχι την ευρώπη του φόβου του σκοταδισμού του περιορισμού των δικαιωμάτων. καλή τύχη στους δικαστές. Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη. Σα ζητώ συγγνώμη γιατί λόγω της μπλε κάρτας ε, πέρασα στο επόμενο βήμα. Και μετά τους ομιλητές από τις ομάδες να ακούσουμε τα μεμονωμένα μέλη και θα δώσω το λόγο λοιπόν στην κυρία Χαλέτσκη. Ένα λεπτό. Κυρία Σίντο, στη δημοκρατία κυρίαρχο είναι το δίκαιο και θα πρέπει να τηρείτε το Σύνταγμα και να μην παραβιάζετε. Κανένα πολιτικό κόμμα, ακόμη και κυβερνό κόμμα, δεν έχει δικαίωμα να παραβιάζει το Σύνταγμα, δεν έχει δικαίωμα να παραβιάζει τις συνθήκες. Γιατί η συζήτηση εδώ δεν αφορά την Πολωνία, αλλά την προστασία του κράτους δικαίου ε, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δικαστές θέλουν να εφαρμόσουν το δίκαιο και να τηρήσουν τις συνθήκες και δεν μπορούν να υφίστανται πειθαρχικέ κυρώσει γι' αυτό και πειθαρχικέ έρευνε. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δράση της. Θα ήθελα ε, να πω και στην πολωνική αντιπροσωπεία του ΕΛΚ ότι φυσικά και είμαι είμαστε υπέρ ενός ψηφίσματος και μιας λύσης που προστατεύει και ενισχύει την Ένωση. Γιατί είμαστε και εμείς πολίτες της Ένωσης και χωρίς ε, κράτος δικαίου δεν υπάρχει ελευθερία. Ευχαριστώ. Danke. Uh, σας ευχαριστώ. έχετε μπλε κάρτα, παρακαλώ. Από τον κύριο Γιάκη. Όχι, ο κύριος Γιάκη είναι στον κατάλογο των ομιλητών. Και εσείς ήσασταν στον κατάλογο των ομιλητών. Πάμε λοιπόν στον επόμενο ομιλητή. Σπουρέκ. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Ε, στην Πολωνία ζούμε το διαρκές καρναβάλι της ε, ε, αποξήλωσης ε, της ε, δικαστικής εξουσίας του συνταγματικού δικαστηρίου. Έχουμε, έργα, έχουμε έλεγχο επί του ορισμού των δικαστών και του ανωτάτου δικαστηρίου. Έχουμε και έναν φημοτικό νόμο που θα δίνει ακόμα λιγότερες δυνατότητες κίνησης εις τους δικαστές. Αυτό αποτελεί κατάφορη παραβίαση του κράτους κράτους δικαίους. Οι δράσεις που έχει αναλάβει η κοινωνία των πολιτών, οι διαμαρτυρίες των δικαστών, καθώς επίσης και η ενεργοποίηση του άρθρου 7 δεν ήρκεσαν. Ε, πρέπει να ε, προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Θα πρέπει ε, να σταματήσουν οι διαδικασίες αυτές στο ανώτατο δικαστήριο και θα πρέπει να βρούμε ένα τρόπο τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην δίνονται σε τέτοιες χώρες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σοφίντβελτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αποφασιστική παρέμβαση ε, που έκανε. Όσον αφορά τους ε, Βρετανούς συναδέλφους του ECR, ε, κοιτάξτε, εσείς δικαιολογείτε αυτήν την κάθαρση το, του, δικαστικού ε, σώματος με περίεργους τρόπους. Αυτό που με εκπλήσει όμως αρνητικά είναι ότι ορισμένοι από τα μέλη της ε, ομάδας σας, ας πούμε το Dutch Forum για τη Δημοκρατία, ε, δεν θέλουν τέτοιου είδους διαδικασίες στην δικιά τους χώρα. Θέλουν ελευθερία και ανεξαρτησία του δικαστικού ε, σώματος και της δικαστικής εξουσίας. Κοιτάξτε, εάν δεν αναγνωρίζετε την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν δεν αναγνωρίζετε την ε, δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, τότε ε, ε, μιλάμε για de facto έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν το λέτε όμως ξεκάθαρα αυτό στους πολίτες ε, της χώρας σας και σε όσους σας ψηφίζουν και στους ψηφοφόρους σας. Πρέπει να είστε ξεκάθαροι. Συνάδελφε, θέλετε, δέχεστε μπλε κάρτα. Από την κυρία Σαλέτσκα. Yes. Κύριε Ζελεύσκα, ευχαριστώ. Κύριε συνάδελφε, χρησιμοποιείτε εκφράσεις που δεν γνωρίζετε, δεν έχετε ιδέα για αυτά που λέτε. Όλοι οι δικαστές στην Πολωνία είναι ελεύθεροι. Η Πολωνία είναι κυρίαρχη χώρα. Πείτε μας, ποια ευρωπαϊκή αξία παραβιάσαμε. Ναι, οι Πολωνοί αγαπούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ναι, θέλουν αλλαγέ και μεταρρυθμίσει στη δικαστική εξουσία. Δώστε μου συγκεκριμένο παράδειγμα. Και κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, όποιο προβουλευτή λαμβάνει το λόγο, να μην μιλάει μόνο με τίτλου εφημερίδων, αλλά να δίνει συγκεκριμένα παραδείγματα. Και τέτοια παραδείγματα δεν υπάρχουν. Κύριε Εντφέλτ, αγαπητέ συνάδελφε, κοιτάξτε. Δεν χρειάζεται να πιστέψετε εμένα προσωπικά, να πιστέψετε ε. του πολλού δικαστέ που κάθονται εδώ πάνω. Και αν ε, δεν ακούτε τους δικαστές ε, που έχουν ορκιστεί στο Πολωνικό Σύνταγμα, μήπως να ακούσετε την ανεξάρτητη γνωμοδότηση και τη δικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αν δεν αναγνωρίζετε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν μπορεί να είστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Στρίκ, τι είναι και. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Την προηγούμενη εβδομάδα οι δικαστές από πάνω από 20 ευρωπαϊκές χώρες ε, μαζεύτηκαν στη Βαρσοβία για να υποστηρίξουν τους Πολωνούς συναδέλφου τους στην ε, ε, προσπάθεια υποστήριξης του δικαστικού σώματος και είναι από τους πολλούς Ευρωπαίους πολίτες που ζητούν να αποταθεί δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη λοιπόν για τους Πολωνούς δικαστές για να σταματήσουν η λειτουργία του πειθαρχικού σώματος. Από ό,τι ξέρουμε όμως αυτή η διαδικασία καλύπτει μία μόνο από τις πολλές απειλές για το πολωνικό κράτος δικαίου. Οι δικαστές από όλο τον κόσμο μιλούν κατά των ε, επικίνδυνων αυτών ε, αλλαγών. Οι δικοί μας όμως ε, ηγέτες σιωπούν. Δεν υπάρχουν τακτικές ανακρίσεις, δεν γίνονται νομικά. Αναλαμβάνονται νομικά μέτρα και όλες αυτές οι αποφάσεις ε, λαμβάνονται χωρίς ομοφωνία. Η ερώτηση λοιπόν προς το Συμβούλιο και προς τα κράτη-μέλη μέσω του Συμβουλίου είναι απλή. Η πολωνική κυβέρνηση πόσο πρέπει να προχωρήσει προτού αρχίσετε ένεργα να προασπίζεστε τις ευρωπαϊκές μας αξίες. Ευχαριστούμε πολύ. Δέχεστε γαλάζια κάρτα. Ναι, τη δέχομαι. Το έδρανο 277. Ερώτηση όμως. Ευχαριστώ. Φαίνεται να γίνεται εδώ πολλοπολωνικός πόλεμος. Μην σας δημιουργηθεί αυτή η εντύπωση. Θα ήθελα να θέσω την ερώτηση και σε συναδέλφους άλλων πολιτικών ομάδων. Πού πήγατε ποιοι ε, δικαστές ε, από τα θεωρία μιλάτε. Μήπως ήταν ε, στις υπηρεσίες ασφαλείας, μήπως ήταν από το πρώην κομμουνιστικό καθεστώς. Πού πήγατε που η αστυνομία, πού ήσασταν όταν η αστυνομία είχε επεβατική συμπεριφορά και επιτέθηκε κατά πολιτών. Πού βρισκόταν τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λέτε ψέματα. Να υπογραμμίσω ξανά ότι εδώ ε, πρέπει να ακούσουμε τις δηλώσεις ε, του Συμβουλίου και της Επιτροπής και να συζητήσουμε τα όσα προστάζει η Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν χρησιμοποιηθεί συγκεκριμένα στοιχεία, συγκεκριμένα γεγονότα και από αυτόν συζητούμε. Και τώρα να πάμε στην απάντηση για την ερώτηση του συναδέλφου και να συνεχιστεί μετά η συζήτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, διότι είναι εντελώς αυθαίρετη η κρίση του συναδέλφου. Αυτό που συζητούμε εδώ είναι οι απειλές κατά του κάτους δικαίου στην Πολωνία. Μια πραγματική δημοκρατία αναγνωρίζει τον διαχωρισμό εξουσιών και ελέγχει του τι είδου έλλειψη ισορροπία μπορεί να υπάρχει. Πρέπει να σεβαστούμε λοιπόν και τι πλειοψηφίε αλλά και τι μειοψηφίε που δημιουργούνται σε μια χώρα. Ε, αυτή είναι μια άλλη απειλή και ελπίζω ότι ο πολωνικό λαό και ιδίω η πολιτική τη Πολωνία θα ε, στραφούν ε, πραγματικά στην ουσία των γεγονότων και του κράτου δικαίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να δουν πού υπάρχουν λήψεις. Ευχαριστούμε ο κύριος Κρά. Συνα... Ε, πρόεδρε, συνάδελφοι. Είμαι δικηγόρος στη Γερμανία. Και βεβαίως, εδώ μιλάμε για τους δικαστές που έχουν ε, να κάνουν και με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο δικαστής είναι ελεύθερος στην κρίση του. Όμως, προς Θεού, αυτό δεν σημαίνει ότι οι ίδιοι οι δικαστές μπορούν να καθορίσουν τις αποφάσεις ή τις διαδικασίες ε, που προβλέπονται από την νομοθεσία. Μιλάμε για μια πολωνική ιδιαιτερότητα. Οι δικαστές μόνοι τους μπορούν να ορίζουν συναδέλφους, προεδρία και σώματα ή διαδόχους. Εδώ το μεγαλύτερο, εδώ πρέπει ο δικαστής να δεσμεύεται μεν από την νομοθεσία, αλλά δεν μπορεί ο ίδιος να αυτοδιορίζεται ή να αυτοελέγχεται. Πρέπει να τηρεί κάποιους κανόνες. Αυτή είναι η διαφορά. Και αυτό ακριβώς συζητούμε. Αυτή είναι η παραβίαση και αυτό είναι το θέμα του κατά πόσον ισχύουν οι παλιοί κανόνες και αν τους σέβεται η πολωνική κυβέρνηση nachdem wir derzeit mehrere επειδή υπάρχουν πολλές γαλάζιες κάρτες και έχουμε ήδη καθυστερήσει θα ήθελα να σας παρακαλέσω να χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό σύστημα για να δηλώσετε ότι επιθυμείτε το λόγο και να μπορέσουμε να δούμε και τη σειρά με την οποία ε, υποβάλλετε το αίτημά σας και να προλάβουμε να υποβάλουμε τις ερωτήσεις όπως δει. Και η συζήτηση να ακολουθήσει την προκαθορισμένη της ε, σειρά. Επόμενος, η κυρία Βυσνιεύσκα. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Η Επίτροπος Γιουρόβα είπε ότι ενθάρρυνε τις πολιτικές αρχές να έρθουν σε επαφή με την Κομισιόν σε ό,τι αφορά τις αλλαγές στο δικαστικό ε, σύστημα στην Πολωνία. Αγαπητέ Επίτροπε, αγαπητή Επίτροπε, μπορώ να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μία ένωση σοβιετικών δημοκρατιών. Είμαστε μία ένωση κρατών μελών με κοινή αποστολή. Είμαστε όμως χωριστές ανεξάρτητες χώρες και θα κρατήσουμε τις αρμοδιότητές μας σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη μας και το δικαστικό μας σύστημα. Εμείς είμαστε μια περήφων, περήφανη, δημοκρατική και ελεύθερη χώρα και δεν μας αξίζει αυτή η συκοφαντία και αυτή η λασπολογία εδώ στο Κοινοβούλιο. Και αυτό γιατί συμβαίνει. Γιατί έχουμε την αντιπολίτευση που έχουμε στην Πολωνία, που στόχος της είναι να αμαυρώσει το όνομα της Πολωνίας στο εξωτερικό. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα παραπληροφόρησης. Ζημίας προς την ίδια του τη χώρα. Στο Κοινοβούλιο έχουμε εδώ διαφορετικά πολιτικά κόμματα και διαφορετικές χώρες. Αλλά κανένα κόμμα αντιπολίτευση δεν φέρεται τόσο άσχημα όσο οι εκπρόσωποι της πλατφόρμας των πολιτών, όπως επωνομάζονται. Κυρίε και κύριοι, περί τίνο πρόκειται. Μπορείτε να βυθομετρήσετε τα πράγματα κι εσείς και να ελέγξετε πόσο μακριά μπορείτε να πάτε, ούτω ώστε να ανακτήσετε και να σφετεριστείτε τις αρμοδιότητες ε, των κρατών μελών. Όταν πάτε πίσω στην, αντιπολί... στην Πολωνία, αγαπητή αντιπολίτευση, πώς θα εξηγήσετε την ε, συμπεριφορά σας. Δέχεστε μία μπλε κάρτα. Ναι. Από την κυρία Λουκεσένσκα. Ναι. Ζητάτε συγκεκριμένα στοιχεία. Δείξτε μου νομοθετήματα, συγκεκριμένους νόμους ε, που αφορούν την μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης που θα βελτιώσουν υποτίθεται τη δικαιοσύνη στην Πολωνία ούτω ώστε η δικαιοσύνη να είναι πραγματικά χωριστή από τις υπόλοιπες εξουσίες και να υπηρετεί τον πολωνικό λαό. Απάντηση. Κοιτάξτε, αν μπορούσατε να διαβάσετε και να καταλάβετε τι διαβάζετε, δεν θα είχατε κάνει καν αυτή την ερώτηση. Σας διαβεβαιώ ότι υπάρχουν άπειρες μεταρρυθμίσεις, τροπολογίες της νομοθεσίας που βελτιώνουν την, ε, νομοθε... την ε, δικαιοσύνη. Στο παρελθόν η δικαιοσύνη ήταν καταπιεστική απέναντι στους πολίτες, έπρεπε να αλλάξει. Εμείς στις εκλογές υποσχεθήκαμε στους εκλογείς μας ότι θα μεταρρυθμίσουμε την ε, δικαιοσύνη και αυτό κάναμε. Υπάρχουν δικαστές οι οποίοι ε, διώκονται γιατί απλώς απαιτούν να εφαρμοστεί το κράτος δικαίου. Ε, υπάρχει δίωξη τη ελευθερία έκφραση, τη ελευθεροτυπία, ε, του δικαιώματο ενημέρωση, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι δραματικό που αυτό συμβαίνει σε μια χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να είμαστε απαιτητικοί και όχι μόνο να ζητήσουμε πολωνική κυβέρνηση να σεβαστεί την Χάρτα Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά και θα πρέπει να μην δεχόμαστε το, τις ρητορίες μίσους της άκρας δεξιάς. Δεν μπορούμε επίσης να δεχτούμε ότι η άκρα δεξιά είναι ένα κανονικό κόμμα όπως τα υπόλοιπα. Αυτά όλα είναι αφηγήματα της άκρας δεξιάς. Ξαναγράφει την ιστορία και ποινικοποιεί την αντιφασιστική δράση και αγώνα. Δεν θέλουμε να δεχτούμε να μας γυρίσετε πίσω σε σκοτεινές εποχές, σε εποχές φασιστικής Ευρώπης. Ο κύριος Γκονζάλες Πόνς. Πρόεδρε, πολύ συγκινήθηκα με ε, την ε, διαμαρτυρία πολωνών δικαστών ε, το προηγούμενο Σάββατο. Ζήταμε να σεβαστεί η κυβέρνηση το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, το Πολωνικό Σύνταγμα, η Ζητάμε οι Πολωνοί δικαστές να σεβαστούν το ευρωπαϊκό δικαστικό σύστημα. Το ίδιο ζητάμε και από κάθε χώρα. Είτε βρίσκεται ανατολικά, δυτικά, βόρεια ή νότια υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα των Πολωνών πολιτών να έχουν ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα. Δεν επιτιθέμεθα στην ε, κυβέρνηση της Πολωνίας. Ε, προστατεύουμε τους ανθρώπους της Πολωνίας, διότι αν πρέπει να διαλέξουμε ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον πολωνικό λαό, πιστέψτε με, ξέρουμε πολύ καλά ποιον θα υπερασπιστούμε. Και ε, συνάδελφοι από το ECR, τώρα ειλικρινά καταλαβαίνετε πόσο βλάπτει η κυβέρνησή σας στη χώρα σας. Συνάδελφε Πόνσε, δέχεστε γαλάζια κάρτα από τον κύριο Τσαλέτσκι. Παρακαλώ, κύριε Τσαλέτσκι. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω ότι οι Πολωνοί πολιτές, που σας ευχαριστώ πολύ που τους αναφέρατε έξι φορές, ε, μας ψήφισαν στις εκλογές. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για την ανησυχία σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή μιλήσατε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι σημαντικό θέμα και για μας. Είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς λοιπόν πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι η χώρα σας απέριψε απόφαση του δικαστηρίου, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όσον αφορά τους καταλανούς ευρωβουλευτές. Κύριε Πόνς. Δύο πράγματα θα πω, ένα στα αγγλικά και ένα στα ισπανικά. Στα αγγλικά ψεύδεστε. Στα ισπανικά ψεύδεστε. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας δέχτηκε την απόφαση του ε, Ανώτατου Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Υπάρχει λοιπόν σημαντική διαφορά. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας ε, σέβεται το δίκαιο. Ψεύδεστε κύριε. Η Καταρίνα Μπάρλη, αντιπρόεδρος, έχει τώρα το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Χθε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ε, ζήτησε ε, αναστολή του μέτρου και ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δράσει γρήγορα. Σήμερα στη Γερουσία συζητιέται το θέμα αυτό, όπου παρεπιπτόντως ε, το κόμμα έχασε την ε, πλειοψηφία. Είδαμε και την εκστρατεία λασπολογίας. Ε, δικαστές διαδήλωσαν στο, στους δρόμους το Σάββατο και εδώ έχουμε θαραλέους ανθρώπους, δικαστές και εισαγγελείς που ήρθαν εδώ στο Στρασβούργο. Από ό,τι καταλαβαίνω, οι άνθρωποι αυτοί δεν θα υποστούν κυρώσεις επειδή συνομίλησαν ε, μαζί μας. Ε, ελπίζω ότι αυτό θα τηρηθεί. Και περιμένω αγωνίως να δω τι θα πείτε στους δικαστές που ήδη ε, έχουν υποστεί κυρώσει διότι θέλουν να εφαρμόσουν το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτό που συμβαίνει στην Πολωνία δεν διαφέρει ε, ε, έχει να κάνει με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Θέλουν να απαγορεύσουν το ευρωπαϊκό δίκαιο. Και έχουμε τον Στάνισλαφ Πρόστοβιτς ο οποίος τη δεκαετία του 1980 έκανε διώξεις ε, υπό το κομμουνιστικό καθεστώς. Ε, μπορείτε σας παρακαλώ να μα τα εξηγήσετε αυτά. Ο κύριος Πάτρικ Γιάκη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μια και είναι τόσο κακό το καθεστώς μας, ε, τι να πούμε για το δικό σας καθεστώ που ε, έλαβε τη μισή υποστήριξη από το δικό μας, αλλά α περάσουμε στην ουσία. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το ότι μιλάτε όλοι με πολύ γενικούς όρους απόψε. Κανείς δεν είπε πώς ε, θεωρεί ότι πολιτικοποιήθηκε η επιλογή δικαστών ε, στην Πολωνία διότι θα μπορούσε να θέσει κανείς και άλλες ερωτήσεις ε, προς την Επίτροπο Γιούροβα. Ε, πώς εκλέγονται οι δικαστές, ε, πώς διορίζονται οι δικαστές στην Τσεχία. Χαίρομαι πολύ που ε, πήρε το λόγο Γερμανός Ευρωβουλευτής. Ε, γνωρίζετε ότι στην Πολωνία δικαστές εκλέγουν άλλους δικαστές. Ε, στη Γερμανία λοιπόν τι γίνεται. Πολύ πρόσφατα μέλος του Bundestag διορίστηκε δικαστής και εσείς έχετε το θράσος να μας μιλάτε για πολιτικοποίηση του δικαστικού συστήματος, κάτι που λέτε ότι δεν ισχύει στην Γερμανία και μιλάτε για την ελευθερία λόγου. είδαμε ε, Γάλλους ε, ε, νομικούς ε, να απορρίπτονται από το, από το εφετείο. Λοιπόν, ε, τώρα πια η Πολωνία δεν κατέχεται από τη Γερμανία. Δεν θέλουμε να δεχτούμε τους μετανάστες που θέλετε να ε, ε, μας επιβάλλετε. Έχουμε λοιπόν την ελευθερία να αποφασίσουμε μόνοι μας τώρα πια. Ευχαριστούμε. Είχα πει ότι θα δεχτώ περιορισμένα αιτήματα με γαλάζια κάρτα. Τώρα έχω μια γαλάζια κάρτα από την κυρία Άννα. Κυρία Ντόναλτ, Χάνα. Κυρία Ντόναλτ. Ευχαριστώ. Κύριε Γιάκη, σας γνωρίζω καλά. Είμαστε φίλοι και συνεργαζόμαστε. Έλα πάμε πάλι στο θέμα της Πολωνίας και συγκεντρωθούμε σε αυτό. Οι Πολωνοί δικαστέ ήρθαν στο ΕΛΚ και μα μίλησαν για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματο στην Πολωνία. Πολλά από όσα έγιναν αντιφάσκουν και με το ευρωπαϊκό δίκαιο όπω έχει αποφανθεί και το ΔΕΚ. Εδώ λοιπόν, τι δημόσιε διαβουλεύσει προηγήθηκαν μέχρι να εγκριθεί το νομοσχέδιο. Βάσει των. Μα είπαν οι δικαστέ, δεν έγιναν καθόλου διαβουλεύσει. Εσείς λοιπόν θα ακολουθήσετε το σύστημα που επιβάλλεται στη χώρα σας ή ό,τι λένε οι δικαστέ, Ευχαριστώ, αλλά δεν ήταν συγκεκριμένα τα στοιχεία που αναφέρατε. Ο συνάδελφος από την Ισπανία είπε ότι ψευδόμαστε. Ε, η ερώτησή μου όμως είναι πότε θα αναλάβει τις ευθύνες του ο καθένας από τη δική του χώρα, όπως ο συνάδελφος από την Ισπανία. Ο κύριος Λένερς. Ο επόμενος από το ΕΛΚ, ο κύριος Λένερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό το Σαββατοκύριακο η εικόνα που είδαμε στη Βαρσοβία ήταν ιστορική. Οι δικαστέ από 27 χώρε κατέβηκαν στου δρόμου για να διαδηλώσουν κατά τη ε, στρέβλωση του κάτους δικαίου. Η κατάσταση έχει φτάσει δραματικέ διαστάσει. Και έτσι υπονομεύεται και υποβαθμίζεται η λειτουργία, το λειτουργήμα το ίδιο και η αναγνώριση των δικαστών σε ένα κράτος όπου θα έπρεπε το σύστημα να είναι ανεξάρτητο ή υπουργό που θέλει να ε, κάνει την ε, δικαιοσύνη υποχείριο του κόμματό τη, δεν μπορεί να αντιταχθεί στην κοινωνία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλει να συνεργάζεται με την ε, χώρα σα, αλλά να μπορεί να την εμπιστευτεί, όπω και τι υπόλοιπε. Έτσι λοιπόν, έχω πλήρη εμπιστοσύνη στι δράσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προστατεύσουμε το κάτω δικαίου και δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε του δικαστέ τη Πολωνία στην τύχη, τύχη του. γιατί το δικό του αγώνα είναι και δικό μα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ζήπελ. Ευχαριστώ. Η δημοκρατία στην Πολωνία κινδυνεύει. Εδώ παρά τις ε, σοβαρές διαμαρτυρίες, ε, το Κοινοβούλιο περιλαμβάνει και άλλα μέτρα αναγκαστικά για τους δικαστές, όπως χρηματικά πρόστιμα ή στέρηση λειτουργήματος. Εδώ λοιπόν όλα αυτά θα μπορούσε κανείς ε, να τα αντιμετωπίσει μόνο με μεγάλη επιφυλακτικότητα. Η συζήτησή μας θα είναι μια από τις πολλές που έγιναν τα τελευταία χρόνια και πραγματικά εδώ αισθάνομαι ότι συνεχώς ε, ότι συνεχώς βλέπουμε το ίδιο εδώ λοιπόν δεν είναι το θέμα μόνο πώς αισθανόμαστε, αλλά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ασχοληθεί με την διαδικασία επί και επισήμως να ενεργοποιήσει τους μηχανισμούς όλα τα απαραίτητα μέσα για δημοκρατική και νόμιμη Ευρώπη. Προτού να είναι πολύ αργά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, συνάδελφε. Και τώρα, κυρία Φιτζέραλτ. Η... Χωρίς τις αξίες μας, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία λόγου ε, και το κράτος δικαίου δεν μπορεί να υπάρξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι αξίες ε, καθοδηγούν τις εργασίε μας εδώ στο Κοινοβούλιο κάθε μέρα και αποτελούν ε, την ουσία που μας κάνει Ευρωπαίους. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε τη συζήτηση αυτή σήμερα, διότι ε, στην Πολωνία δυστυχώς ε, κινδυνεύουν αυτές οι αξίες. Πρέπει να αναλυφθεί η δράση για να αλλάξει η κατάσταση κατάσταση, ε, διότι με τη διαδικασία του άρθρου 7 ε, πολύ λίγη πρόοδος έχει σημειωθεί. Ελπίζω η πολωνική κυβέρνηση να αλλάξει η πορεία και να σέβεται το δικαστικό σύστημα όπως περιγράφεται στις συστάσεις ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Δεκεμβρίου. Ε, καλό λοιπόν την κυβέρνηση να το κάνει αυτό και να σταματήσει την πολιτική άρνηση που βλέπουμε εδώ σήμερα. Αν δεν γίνει αυτό όμω, θα πρέπει να ε, ε, προχωρήσει η διαδικασία του άρθρου 7. Ε, δεν ε, μπορούμε να δεχτούμε άλλη καθυστέρηση και ε, συμφωνώ με τους νομικούς σε όλους στην Ευρώπη που βλέπουν την αδικία και υπερασπίζονται το κράτος δικαίου που αξίζει τον κόπο να υπερασπιστούμε. Ευχαριστώ. Σιμωσέιβιτς, παρακαλώ. Η κυβέρνηση και το, κρατικό, και το κόμμα στην εξουσία ε, παραβιάζει το κράτος δικαίου. Ε, το Δεκέμβριο ε, με ένα νομοσχέδιο τιμωρούνται οι δικαστές οι οποίοι εφαρμόζουν τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο δεν θα υπάρχει ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Ο πρόεδρος της Γερουσίας που ήρθε στις Βρυξέλλες για να συζητήσει με την κυρία Βέρα Γιούροβα κατηγορείται από την κυβέρνηση ότι υποσκάπτει τα συμφέροντα της Πολωνίας. Και κατηγορείται για παράνομες ε, και αντισυνταγματικές δραστηριότητες. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ε, το κράτος δικαίου, αλλά και τα δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες. Η κατάσταση απαιτεί ε, επίγουσα δράση από το Κοινοβούλιο, την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Είναι θέμα αξιοπιστίας αυτών των θεσμικών οργάνων. Ο κύριος Πόσπισιλ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Θα αναφερθώ σε αυτό που είπε ο κύριος Γιάκη, που μίλησε για το, τη δικαιοσύνη στην Τσεχία. Εγώ ήμουνα υπουργό Δικαιοσύνης της Τσεχίας και ήμουνα υπεύθυνο για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, γιατί είχαμε αντίστοιχα προβλήματα με τους δικαστές στην Τσεχία. Αλλά ποτέ σε καμία περίπτωση δεν μειώσαμε τον πύχη ε, του συνταξιδοτικού ορίου, δεν κατεβάσαμε το συνταξιδοτικό όριο δηλαδή. Παρότι είχαμε παρόμοια προβλήματα. Επομένως, μην ε, περιφρονείτε την ε, τσεχική δημοκρατία που προσπαθήσαμε να κάνουμε τις σωστές μεταρρυθμίσεις με βάση το κράτος δικαίου. Κυρία Γιούροβα, έχετε μια δύσκολη κατάσταση στα χέρια σας και προσεύχομαι ούτω ώστε να πείσετε την Πολωνική Βουλή, ούτω ώστε να κάνει τι μεταρρυθμίσει στη μετακομμουνιστική περίοδο με σεβασμό του κράτου δικαίου. Εμεί αυτό το κάναμε στην Τσεχία και είναι η σειρά σα να στηρίξετε το κράτο δικαίου και παράλληλα να έχετε μία μη κομμουνιστική δικαιοσύνη. Ευχαριστώ. Μπιεντρών. Ευχαριστώ. Έχω άσχημα νέα για σας. Τα δικαστήρια είναι ακόμα ζωντανά, όπως όσο ζωντανοί είμαστε κι εμείς. Προσπαθείτε να μας φημώσετε, αλλά η πολωνική κοινωνία θα κατεβαίνει στους δρόμους όσο χρειάζεται για να υπερασπιστεί το Σύνταγμα και το κράτος δικαίου και την συνταγματική τάξη της χώρας θα συνεχίσουμε να δείχνουμε αλληλεγγύη και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τον πολωνικό λαό. Γιατί εσείς, οι δικές σας ελίτ, αποτελούν απειλή για το κράτος δικαίου στην Πολωνία και για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας προειδοποιώ λοιπόν τώρα. Εάν συνεχίσετε σε αυτή την άγουσα, θα βρεθείτε ακόμα πιο απομονωμένοι θα φτάσετε κοντά στη Ρωσία, εκεί μαζί με τη Λευκορωσία. Θα έχετε τους ίδιους καονισμούς, όπως αυτές τις χώρες. Συνέχεια μιλάτε για τις ελίτ. Ποιες είναι αυτές οι ελίτ τώρα στην Πολωνία, εσείς είσαστε αυτές οι, οι νέες ελίτ. Μία νεοκομμουνιστική ελίτ στην Πολωνία. Ελέγχετε τα ΜΜΕ, ελέγχετε τη Βουλή, ελέγχετε τον πρόεδρο. Είσαστε δηλαδή, είναι ο πρώτος σας τα δικαστήρια. Επομένω, προσοχή, δεν θα σπάσετε ποτέ την αλληλεγγύη μα. Ευχαριστώ. Επόμενο ομιλητή, ο κύριο Μουρεσάν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Ρουμάνος είμαι και η προηγούμενη κυβέρνηση της Ρουμανίας προσπάθησε να αποδυναμώσει το δικαστικό σύστημα και ε, το κράτος δικαίου. Και είδαμε πώς, πόσο αποφασιστικά οι πολίτες διαδήλωσαν στους δρόμους με ευρωπαϊκές σημαίες στα χέρια τους ε, περιμένοντας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα να σταθούν στο πλευρό τους. Ε, και τι έγινε. Ε, οργανώθηκε δημοψήφισμα από τον Πρόεδρο και ήταν σαφές το αποτέλεσμα. Πάνω από το 85% των ανθρώπων είπαν ότι θέλουμε ισχυρό δικαστικό σύστημα. Δεν θέλουμε αδιαφανείς αλλαγές στο σύστημα αυτό. Ε, ούτε θέλουμε να εφαρμοστεί μαζική αμνηστία. Και γι' αυτό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ στο Στρασβούργο λέω στου ανθρώπους της Πολωνίας «Ε, σας ακούμε, σας υπερασπιζόμαστε και το ίδιο λέω και στους δικαστές της Πολωνίας. Είναι καθήκον μα να σα υπερασπιστούμε και τις ευρωπαϊκές αξίες σε κάθε γωνιά της Ευρώπη. Κάθε προσπάθεια αποδυνάμωσης του δικαστικού συστήματο ε, ε, είναι απαράδεκτη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αγωνιστεί γι' αυτό. Ευχαριστώ. Η κυρία Τούν Χόνσταϊν. Έχετε γαλάζια κάρτα? Κύριε Μουρεσάντα, έχετε τη γαλάζια κάρτα? Ναι, τη δέχομαι, διότι θέλω να μιλήσω περισσότερο, ναι. Κυρία Τούν Χόινστάιν, παρακαλώ. Συνάδελφε, Μιλήσατε με σαφήνεια και έχω μια ερώτηση προς εσάς. Θέλω να σας ρωτήσω. Εσείς πώς ε, βλέπετε την χρήση πειθαρχικών κυρώσεων ε, σε βάρος των δικαστών. Ε, ένα παράδειγμα να σας δώσω. Ένας, παρόν είναι, ένας από τους δικαστές είναι παρόν και 55 πειθαρχικές διαδικασίες έχουν ξεκινήσει κατά του ε, για εφαρμογή αποφάσεων ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Εσείς πώς βλέπετε αυτές τις διαδικασίες. Ο κύριος Μωρεσάν, ευχαριστώ συνάδελφε για την ερώτησή σας. Όποτε ε, ε, οι πολιτικοί θέλουν να συγκεντρώσουν όλη την εξουσία, ε, επιτίθενται στην αντιπολίτευση, στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη και θα επιτίθενται σε δικαστές υπό τον ελεγχό τους. Πάντα είναι κακό σημάδι όταν οι κυβερνήσεις θέλουν να περιορίσουν τις δυνατότητες της δικαιοσύνης. Ποτέ δεν θα πρέπει η δικαιοσύνη να υπακούει στην κυβέρνηση, είναι ανεξάρτητη εξουσία και έτσι θα πρέπει να παραμείνει. Σας ευχαριστώ πολύ. Προχωράμε στη διαδικασία Catch the Eye. παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι Είδαμε τι ακριβώς κάνει η κυβέρνηση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην εξουσία στην Πολωνία. Αλλά η συζήτηση αυτή δεν αφορά την Πολωνία, αφορά το μέλλον τη Ευρώπης, την ασφάλεια των παιδιών μας. Ε, ε, ε, αν επιτρέψουμε, αν ανομία σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης, αυτό θα είναι δική μας ευθύνη, δικό μας θέξιμο. Εάν οι δικαστές ε, που δεν επιθυμούν να υπακούσουν ε, στους ε, κομματάρχες, αυτό θα αποτελέσει δική μας ευθύνη. Εάν επιτρέψουμε να τιμωρούνται οι αθώοι, θα είναι δικό μας το φταίξιμο. Εάν επιτρέψουμε στην προπαγάνδα αυτή να μας πλημμυρίσει, δική μας αποτυχία θα είναι. Μερικοί λένε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι ε, συνεργάτες του κυρίου Πούτιν, ε, αλλά δεν ε, μιλάμε για ομάδα, μιλάμε για χιονοστιβάδα. Ευχαριστούμε. Περνάμε τώρα στη δικασία Catch Έχουμε πολλές παρεμβάσεις. Θα κοιτάξω να πάρω από κάθε πολιτική ομάδα έναν αγορητή. Ξεκινάμε με τον κύριο Τσεχόφκη. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, συνάδελφοι. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι είμαι προκατελημένος κατά της Πολωνίας. Είμαι μεγάλος φίλος της Πολωνίας και ανέκαθεν προασπιζόμουν την φιλία Τσεχίας-Πολωνίας. Ωστόσο, όταν ανέγνωσα το σχέδιο ε, το, σχέδιο, το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, πραγματικά ανατρίχιασα. Δεν θέλω να καταδικάσω την Πολωνία, δεν θέλω να επικρίνω κανέναν, πάντοτε σας υπερασπιζόμουν. Όμως, ας αξιοποιήσουμε τη συζήτηση αυτή, όχι για να τσακωθούμε μεταξύ μας, αλλά για να καθίσουμε γύρω από το ίδιο τραπέζι και να κοιτάξουμε να αρχίσουμε συζήτηση για τη μεταρρύθμιση αυτή. Το θέμα δεν είναι να επικρίνουμε κανέναν. Απλώς θέλουμε να πούμε ξεκάθαρα ότι κάποια από τα βήματα, κάποια από τα σημεία της μεταρρύθμισής σας πάνε πολύ μακριά. Πράγματα που δεν έχουν συμβεί λόγω χάρη ποτέ στη Δημοκρατία της Τσεχίας. Ευχαριστούμε ο κύριος Μπενχαμπή. Κυρίες και κύριοι, η Πολωνία είναι ένα από τα μεγαλύτερα έθνη στην Ευρώπη και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει μακρά ιστορία δημοκρατίας και μάλιστα ε, μια μορφή δημοκρατίας υπήρχε στη χώρα πρωτού από πρώτα, πριν από κάθε άλλο κράτος ή χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Πολωνία 45 χρόνια αγωνίστηκε για την ελευθερία της ε, κατά της έσου Εδώ λοιπόν δεν μιλάμε για κάποιο σώμα που μόνο του έχει ορίσει ε, κάποιο πολιτικό σώμα. Ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει 28 διορισμένους δικαστές. Δεν μιλάμε για κάποιο σώμα που έχει μια κυβέρνηση σαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την οποία δεν έχει κλέξει κανείς. Πώς μπορούμε να κατηγορούμε ένα πολιτικό κόμμα που έχει εκλεγεί δύο φορές και έχει κληθεί να κυβερνήσει τη χώρα ε, και μάλιστα να χρησιμοποιούμε ως μανιφέστο εναντίον του τη μεταρρύθμιση του δικαστικού σώματος. Πραγματικά αυτό που έχω να πω σε εσά που κυβερνάτε είναι να μην ανεχτείτε αυτέ τι πιέσει. Θα βρείτε φίλου στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα σα στηρίξουμε. Και... Ευχαριστούμε. Η Μπεάτα Κέμπα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Μπιεντρών, μιλάτε για Ρωσία και Λευκορωσία. Οι χώρες αυτές έχουν τις δικές τους αξίες και ε, χρειάζεται να υποστηρίξουμε και με αυτέ τη συνεργασία μα ε, η μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος. Ακούσαμε τι είπε η Επίτροπο Γιούροβα. Τι θα γίνει με το διορισμό των δικαστών όμως. θα μιλήσετε ατομικός, προσωπικός, με όσου αν υποτίθεται. για τα θέματα του δικαστηρίου. Ο δικαστής γνωρίζει πολύ καλά τι κάνει. Εσείς όμως τι ακριβώς θέλετε, διότι και εγώ η ίδια αισθάνομαι ότι φύγομαι. Και σίγουρα είναι ανησυχητικό αυτό. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε να βάλουμε φωτιά στο δικό μας το σπίτι. Ε, Αυτά είχα να πω, κυρία Επίτροπε. Ευχαριστούμε, συνάδελφε. Ο κύριος Ντούντα δεν είναι εδώ, οπότε λίγη η συζήτηση και θα ακούσουμε την εκπρόσωπο της τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Ρέιντερς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να απαντήσω σε κάποια θέματα που ακούστηκαν για το κράτος δικαίου στην Πολωνία. Θέλω να επανέλθουμε στην χθεσινή απόφαση του Σώματος των Επιτρόπων να ζητήσουν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να πάρει μέτρα στα πλαίσια των διαδικασιών που είναι εξελίξει για να αναστείλει τη λειτουργία του πειθαρχικού σώματος ε, στην Πολωνία. Όπω είπε και η κυρία Γιούρεβα, παρά την ε, προδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, τα, οι, δικαστές των τακτικών δικαστηρίων που προσπαθούν να εφαρμόσουν αυτή την απόφαση υπόκεινται πειθαρχικέ διαδικασίε και το πειθαρχικό σώμα εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικότατα. Λόγω του κινδύνου που υπάρχει για φοβερή βλάβη εναντίον των δικαστών στην Πολωνία, Ήδη το Δεκέμβριο ήρθα σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές στην Πολωνία για να παρακολουθούν εκ του σύνεγγες την κατάσταση, ούτω ώστε να πάρει και το σώμα των επιτρόπων τι σωστέ αποφάσεις και τις πήραμε χθε. Ενδιάμεσε αποφάσεις. Χρειαζόταν να γίνει κάτι τέτοιο, ήταν επίγον. Σε ό,τι αφορά το νέο νομοσχέδιο που είναι στα τώρα στα σκαριά και στα πλαίσια της νομοθετικής διαδικασίας. Η Επιτροπή της ε, Βενετίας θα πάρει μια απόφαση. Θα πρέπει οι συστάσεις της Επιτροπής της ε, Βενετίας να εφαρμοστούν πλήρως στα πλαίσια της νομοθετικής διαδικασίας. Η Κομισιόν εκαλεί τις πολωνικές αρχές να μην προωθήσουν, να, να μην προχωρήσουν με αυτό το νέο νομοσχέδιο πριν κάνουν όλες τις απαραίτητες διαβουλεύσεις. Η γνώμη της Επιτροπής ε, της Βενετίας θα ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση που θα κάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άκουσα εκκλήσει για ένα νέο μηχανισμό για το κράτο δικαίου. Σας διαβεβαιώ ότι η Κομισιόν θα εργαστεί για να υπάρξει ένας ευρύς μηχανισμός για το κράτο δικαίου, κατά προτεραιότητα, θα καλύπτει όλα τα κράτη-μέλη και θα λάβει υπόψη τις διάφορες συνιστώσεις του κράτους δικαίου, Φερρυπίν, ε, θα λαμβάνει υπόψη τα συστημικά προβλήματα ε, για το πώς ενεργοποιούνται διάφοροι νόμοι, πώς περνάνε δηλαδή από τη Βουλή οι νόμοι, τι κάνουν ε, τα δικαστήρια, είναι ανεξάρτητα τη δυνατότητα καταπολέμησης της διαφθοράς και τον πλουραλισμό των ΜΜΕ. Θα προσπαθούμε να εντοπίζουμε εγκαίρως τα προβλήματα που υπάρχουν σε επίπεδο κράτος δικαίου. Μετά από κάποιες παρατηρήσεις που άκουσα, θέλω να σας πω ότι κάθε δικαστικό σύστημα είναι διαφορετικό και θα πρέπει να το εξετάζουμε πάντα με ένα πλήρη και συνεκτικό τρόπο. Δεν μπορούμε να απομονώνουμε μία συγκεκριμένη διάταξη ενός κράτους μέλους και να το συγκρίνουμε με μία άλλη μεμονωμένη διάταξη ενός άλλου κράτους μέλους, χωρίς να κοιτάμε το πλαίσιο του δικαστικού συστήματος και της ένομης τάξης καθώς και των επιπέδων ελέγχου που υπάρχουν σε κάθε κρατός μέλος. Όπως είπε και στην αποφασή του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η οργάνωση της δικαιοσύνης στα κράτη-μέλη είναι αρμοδιότητα των ιδίων των κρατών μελών. Παραμένει γεγονός ότι όταν ασκούν αυτές τις αρμοδιότητες τα κράτη-μέλη, πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο. Το κράτος δικαίου είναι το θεμέλιό μας. Και δεν πρέπει να υπάρξουν συμβιβασμοί εκεί. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι γίνεται σεβαστό το κράτος δικαίου και στηρίζεται πάντα. Κλείνοντα, Πρόεδρε, η Κομισιόν θα συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση στην Πολωνία εκ του Σύνεγγυ. Και θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε επικοδομητικό διάλογο με τι πολωνικέ αρχέ. Η εισαγωγή τη διαδικασία επιπαραβάση δεν αποκλείει το διάλογο θα είμαι στο Ζάγκρεπ, στην άτυπη Υπουργική Σύνοδο των Υπουργών ε, Δικαιοσύνης, 23 και 24 Ιανουαρίου. Καλό τον Πολωνό Υπουργό Δικαιοσύνης να υποφεληθεί από αυτή την ευκαιρία, από αυτή τη συνάντηση και να συνομιλήσει μαζί μου επικοδομητικά. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, περιμένουμε με αγωνία την απάντηση του Συμβουλίου. Κύριε Μπερνάκης, παρακαλώ. Σας διαβεβαιώ ότι η Προεδρία και το Συμβούλιο ε, το συνόλο του δίνει μεγάλη σημασία σε αυτό το θέμα. Πιστεύουμε ότι μόνο μια κοινή προσπάθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσμούς της, καθώς και τα κράτη-μέλη, θα επιτρέψουν στην Ένωση να εξασφαλίσουν ότι το κράτος δικαίου είναι ο κρογωνιαίος λήθος του κοινού μας εγχειρήματο. Το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων συζήτησε αυτό το θέμα της Πολωνίας τα τελευταία δύο